Good uh, Καλησπέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι και κύριες και κύριοι. Συνεχίζεται η σύνοδος. Τα πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης και τα εγκεκριθέντα κείμενα έχουν ήδη μοιραστεί. Αν δεν υπάρχουν σχόλια, εγκρίνονται τα πρακτικά. Και μπορούμε να περάσουμε στο πρώτο σημείο της ημέρησης διάταξής μας, που είναι η συζήτηση επικαιρότητα για την ε, έκτακτη ανάγκη στα θέματα του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής. Δεν θα γίνουν δεκτές ερωτήσεις με τη διαδικασία της μπλε Θα ήθελα να δώσω το λόγο τώρα στην πρώτη ομιλήτρια, την κυρία Ντάλη. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τους συναδέλφους που είναι παρόντες στη συζήτηση. Ευχαριστώ την εκπρόσωπο της Φιλανδικής Προεδρίας. Ελπίζω ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμερίζεται την επιτεκτική ανάγκη που είναι η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και να έρθει και ο εκπρόσωπος. ανεβαίνει η σταθμή της θάλασσας και επίπεδα που γίνονται μία φορά το αιώνα κανονικά αναμένονται να γίνονται μία φορά το χρόνο μέχρι το 2050 σε πολλές διαφορετικές μέρες και η πυρκαγιές ε, των δασών φαίνεται θα αυξηθούν μέχρι τα τέλη του αιώνα και δεν είναι δικές μου δηλώσεις. Είναι μερικά από τα συμπεράσματα της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπως προκύπτουν από την τελευταία έκθεση του Σεπτεμβρίου. Η κλιματική αλλαγή, η κλιματική κρίση και η κατεπίγουσα ανάγκη στα θέματα αυτά έχει απασχολήσει τους πάντες και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε επιδύσει από τα κενά λόγια εκείνων που λένε ότι η κλιματική αλλαγή θα πρέπει να αντιμετωπιστεί κατεπηγόντως, αλλά από την άλλη όταν πρέπει να λάβω μέτρα δεν δείχνουν την ίδια τόλμη. Θα πρέπει να συζητήσουμε κάποια μέτρα που θα κάνουν τη διαφορά. Γιατί οι πολίτες πληρώνουν τα σπασμένα των πυρκαγιών, των καταιγίδων και των ε, πλημμυρών. Θα πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε τα αίτια αυτού του κακού που οδηγεί σε ακραία καιρικά φαινόμενα και γι' αυτό και οι σοσιαλιστέ δημοκράτε ζήτησαν τη διοργάνωση τη συζήτηση. Θέλουμε μια νέα προσέγγιση να αντιμετωπίσουμε αυτή την έκτακτη ανάγκη του κλίματο. Γιατί πρόκειται για έκτακτη ανάγκη. Και μπορεί να θεωρούμε ότι είναι έκτακτη ανάγκη και κατεπίγουση κατάσταση. Δεν αρκεί να το δηλώνουμε. Γιατί όταν καίγεται το σπίτι σου, δεν πατά απλώ στο συναγερμό και κάθεσαι με σταυρωμένα χέρια θα πρέπει να έρθει το πυροσβεστικό και να κατασβεστεί η πυρκαγιά στο σπίτι σου. Γι' αυτό και εμεί θα πρέπει να αρχίσουμε τώρα τι εργασίε. με ένα μακροπρόθεσμο κοινωνικό και περιβαλλοντικό σχέδιο, με νομοθετικέ προτάσει ε, που θα συνοδεύονται από κατάλληλε επενδύσει και σωστή εφαρμογή. Χρειαζόμαστε χρήματα για να χρηματοδοτήσουμε την απαιτούμενη μετάβαση το συντομότερο δυνατό από, από τον επόμενο χρόνο. Χρειαζόμαστε και δημόσια και ιδιωτικά κονδύλια σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Για την ουδετερότητα του, θα, άνθρακα θέλουμε ρηξικέλευθες μεταρρυθμίσεις για να δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης και να εξασφαλίσουμε τη βιομηχανική μας ανταγωνιστικότητα, την αθεκτικότητα ε, των επιχειρήσεών μας και να βελτιώσουμε την ποιότητα και την ανθρώπινη υγεία. Επίσης, θα πρέπει να απαλλαγούμε σύντομα από τις εκπομπές άνθρακα και θα πρέπει να μετα... να απομακρυνθούμε από τα ρηκτά καύσιμα προς πιο φιλοπεριβαλλοντικέ τεχνολογίε με καθαρή παραγωγή ενέργεια, στηρίζοντα τη βιοπικιλότητα και αναπτύσσοντας ένα νέο αηφόρο γεωργικό μοντέλο για να αποφύγουμε την ε, ε, έλλειψη τροφίμων. Επίση, θέλουμε κατάλληλα σχέδια αναδάσωσης ή δάσωση περιοχών. Επίσης, ε, να αναπτύξουμε νέε τεχνολογίε για να αντιμετωπίσουμε τη λειψιδρία. Θέλουμε καινοτομία και να εξασφαλίσουμε ε, νέα και πιο ε, ενεργειακά αποδοτικά κτίρια με σωστή ανακαίνιση των προηγούμενων κτίριων. Επίσης θέλουμε αυτό να γίνεται χωρίς να αφήνουμε κανένα πίσω, με κοινωνική πρόοδο. Θέλουμε λοιπόν μια κλιματική δράση που θα επιτύχει το 21% των απαραίτητων μειώσεων εκπομπών μέχρι το 2050. Επίσης, ε, θέλουμε παραγωγή ενέργειας που θα στηρίζεται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θα πρέπει να αναπτύξουμε εναλλακτικά καύσιμα ε, και να προστατεύσουμε τα θαλάσσια οικοσυστήματα και τι ε, πηγέ τροφίμων που βρίσκονται στου ωκεανού. Υπάρχει όλο και μεγαλύτερη επαγρύπνηση και συνειδητοποίηση. Οι νέοι έχουν αρθρώσει λόγο και θα πρέπει να κάνουμε μια επιλογή. Ήδη απλώ να δηλώνουμε ότι έχουμε κρίση και να μην κάνουμε τίποτα αυτό και συγκεκριμένο ή να χρησιμοποιήσουμε αυτή την πρόκληση για να ενισχυθούμε και να ενδυναμωθούμε. Εμείς ε, όσοι σοσιαλιστές και δημοκράτες επιλέγουμε τη δεύτερη λύση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ και τώρα εκ μέρους... Εκ... Ευχαριστούμε της Φιλανδικής Προεδρίας, κυρία Τουπουρένεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που με προσκαλέσατε για να εκπροσωπήσω το Συμβούλιο σε αυτή την τόσο σοβαρή συζήτηση την κέρια σημασία συζήτηση. Έχει γίνει υπαρξιακή απειλή ε, από την οποία δεν απαλλάσσεται και δεν γλιτώνει καμία χώρα. Πρέπει όλοι να προσέξουμε για τις επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών και πρέπει να επιτείνουμε τις προσπάθειές μας. Να χρησιμοποιήσουμε τα προσφατότερα επιστημονικά στοιχεία ε, και να αξιοποιήσουμε όλα τα περιβαλλοντικά πάνελ για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών έχουμε 1,5 βαθμό αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας σε, σχέση με τα επίπεδα πριν τη βιομηχανική επανάσταση. Ήδη η υπερθέρμανση του πλανήτη έχει περάσει τον 1 βαθμό ε, και θα φτάσει τους 0,2 βαθμούς αύξηση ανά δεκαετία. Εάν δεν ε, εντείνουμε τις ε, παγκόσμιες προσπάθειές μας, μπορεί να φτάσουμε την αύξηση πάνω από 2 ε, βαθμούς Κελσίου μετά το 2060 και αυτό θα συνεχιστεί και μετά. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τον αλληλοσχετισμό με τη βιοποικιλότητα, τους υδάτινους πόρους και τα οικοσυστήματα. Η Αρκτική ε, υπερθερμαίνεται διπλάσια σε σχέση με τον υπόλοιπο πλανήτη και αυτό έχει παγκόσμιες και τοπικές συνέπειες. Όμως, ε, βάσει των μελετών του ΟΗΕ, οι εθνικές συνεισφορές που έχουν ε, υποβάλει τα μέρη της Συμφωνίας των Παρισίων δείχνουν ότι καθυστερούμε για την επίτευξη των μακροπόθεσμων στόχων της Συμφωνίας. Και παρόλο που δεν έχει γίνει ως τώρα επαρκής πρόοδος, χρειάζεται περισσότερη ε, φιλόδοξη δράση με εντονότερο ρυθμό. Υπάρχουν θετικά δείγματα ότι υπάρχουν περισσότερε γνώσει, ενημέρωση και ανησυχία για τι κλιματικέ αλλαγέ και τι επιπτώσει του ε, σε όλο τον κόσμο. Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό να βλέπουμε ότι η κοινωνία των πολιτών και οι πολίτε, ιδιαίτερα οι νέοι, καλούν για περισσότερη και πιο φιλόδοξη δράση. Οι ανθρωπογενείς ε, ρήπανση που προκαλείται, σχετίζεται με τις κλιματικές αλλαγές και έχει φτάσει σε αυτήν την αλλαγή του περιβάλλοντος σε σχέση με τις προβιομηχανικές περιόδους, επηρεάζει κυρίως τους νέους. Αυτοί θέλουν να βεβαιωθούν πάνω από όλου ότι θα έχουν ένα πλανήτη στον οποίο θα μπορούν να ζήσουν εκείνοι και μελλοντικέ γενναίες. Η Σύνοδος για το Κλίμα τον περασμένο μήνα ήταν άλλη μια ευπρόσδεκτη πρωτοβουλία για να εντείνουμε τις συλλογικές μας προσπάθειες προς την επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας των Παρισίων η κοινή αυτή συνέστηση και η κοινή βούληση μεταξύ κυβερνήσεων, πολιτών και επιχειρήσεων είναι αυτό που χρειαζόμαστε για να πετύχουμε αλλαγή μοντέλου και να μετατρέψουμε τις, οικονομί, τις οικονομίες μας και τις κοινωνίες μας για να αντιμετωπίσουμε τις βλαβερές συνέπειες των κλιματικών αλλαγών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αποφασισμένη να έχει περισσότερη και πιο φιλόδοξη δράση και θα συνεχίσει να αποσυνδέει την οικονομική της ανάπτυξη από τις εκπομπές ε, αερίων του θερμοκηπίου και από το 1990 στο 2017 είχαμε αύξηση 58% ενώ συνολικά οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μειώθηκαν κατά 22% η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πετύχει τους στόχους της ε, για την μείωση των αερίων του θερμοκηπίου ως ε, το 2020 και μάλιστα με το παραπάνω. Υπάρχει ένα πλήρες νομοθετικό πακέτο που λειτουργεί γιατί έχουμε και νέους στόχους για το 2030 και θέλουμε ε, να, κάνουμε, να αναλάβουμε το δικό μας μερίδιο ευθύνη στη Συμφωνία των Παρισίων όπως δεσμευτήκαμε. Ξέρουμε όμως ότι οι σημερινές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα είναι αρκετές αν δούμε την κλίμακα των μειώσεων που απαιτούνται για να πετύχουμε τους μακροπρόθεσμους μου στόχου μείωση τη συμφωνία. Γι' αυτό γοργή και ε, βαθιά αλλαγή στην κοινωνία και στην οικονομία είναι κάτι είναι μια προπόθεση για τι ερχόμενε δεκαετίε. Εδώ θα πρέπει όλοι να συμμετέχουν και η Ευρωπαϊκή Ένωση να υποβάλει μια μακρόπνοη στρατηγική ε, στα πλαίσιο του πάνελ του ΟΗΕ για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών μέχρι το 2030. Για να προετοιμαστούμε για αυτή την ε, μακροπρόθεσμη στρατηγική, συζητούμε στο Συμβούλιο από τον περασμένο Νοέμβριο πώ θα πετύχουμε την κλιματική ουδετερότητα βάσει τη Συμφωνία των Παρισίων και του μακροπρόθεσμου προγράμματο τη Επιτροπή Ένα καθαρό πλανήτη για όλου, Clean Planet for All. Χρειάζεται μετατροπή στην οικονομία και την κοινωνία για να μπορέσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση όλοι οι τομεί να έχουμε αύξηση των προσπαθειών μα και να πετύχουμε το στόχο μας. Χρειάζεται μια συμμετοχική, ευρεία και εκτεταμένη συγκέντρωση προσπαθειών όλων των κρατών μελών. Η μετάβαση αυτή θα επηρεάσει τους πάντες. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε ότι είναι δίκαια και κοινωνικά ε, σωστά εξισορροπημένη για όλους τους πολίτες. Πρέπει να λάβουμε υπόψη τις ιδιαιτερότητες των κρατών μελών και των διαφορετικών περιοχών και να βεβαιωθούμε ότι κανείς δεν θα μείνει πίσω. Ε, από την άλλη, η μετάβαση αυτή ε, προσφέρει και νέε πράσινε ευκαιρίε καθώ και δυνατότητε για οικονομική ανάπτυξη, νέε θέσει εργασία και τεχνολογική ανάπτυξη. Για να μπορέσουμε να κάνουμε πράξη αυτό το δυναμικό, χρειάζονται ερευνέ που θα πρέπει να ενταθούν ε, με γοργότερου ρυθμού να προστατεύσουμε την τεχνολογία μα από τι διεθνεί πιέσει στο ε, παγκόσμιο προσκήνιο. Τα περισσότερα κράτη-μέλη συμφωνούν με το στόχο τη κλιματική ουδετερότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση το 2050 και πολλά κράτη-μέλη ήδη έχουν προβλέψει εθνικού στόχου για να συνεισφέρουν προ το στόχο. Είμαστε αποφασισμένοι να εργαστούμε επί μια συμφωνία στην οποία θα δεσμευτούν όλα τα κράτη-μέλη και ελπίζουμε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα ε, ολοκληρώσει τι κατευθυντήρε γραμμέ τη για την μακροπρόθεσμη κλιματική στρατηγική πριν το τέλο του 2019. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Και τώρα εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Επίτροπο Έτιγκερ. Παρακαλώ. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι βουλευτέ, κύριε και κύριοι, αξιότιμη προεδρεύουσα πρόσωπε του Συμβουλίου. Ε, εγώ εκπρόσωπο τον συνάδελφο ε, που είναι αρμόδιος για αυτά τα θέματα εξ ονόμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σωστά. Η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ε, δηλώσει ως προτεραιότητα την προστασία του κλίματος, του περιβάλλοντος και γενικότερα του πλανήτη. Υπάρχει μια προεργασία στο προηγούμενο κοινοβούλιο και στην Επιτροπή Juncker και μπορούμε να βασιστούμε. Δεν είμαστε στην αρχή του εξευρωπαϊσμού της αηφορίας και της βιωσιμότητας της πολιτικής κλίματος με κοινά μέσα εργαλεία και δυνατότητες. Στην παγκόσμια σκηνή μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η Ευρώπη έχει αποδείξει φιλοδοξίες και πριν τη Συμφωνία του Παρισιού και μετά τη Συμφωνία του Παρισιού. Και η τήρηση των στόχων είναι δεδομένη για μας. Θα παραμείνουμε κάτω των δύο βαθμών ε, θέρμασης, για να μην πω κάτω του 1,5 βαθμού που θα ήταν το ιδεώδες. Σε αυτό δεν συμφωνούν όλοι παγκοσμίω ε, στη συζήτηση. Έχει νόημα επίσης όλα αυτά να τα αντιμετωπίσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι' αυτό θεωρούμε ότι είναι η δεύτερη καλύτερη λύση ε, ένας μεμονωμένος εθνικός δρόμος του κάθε κράτους μέλους. Νόημα ε, έχει όταν γίνεται αυτό σε μεγαλύτερη κλίμακα, σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Γι' αυτό έχουμε το σύστημα εμπορίας εκπομπών ρήπων, ETS, που με τη μείωση των ρήπων, του όγκου των ρήπων, είναι κάτι που μας ε, απασχολεί και το εξετάζουμε και μπορεί να το αλλάζει ε, κανείς με όρους οικονομίας της αγοράς. Και μέχρι το 2020-2030 θα έχουμε μειώσει ε, μέχρι 50% και μέχρι το 2050 μπορούμε να λειτουργούμε ουδέτερα προς το κλίμα. Λειτουργεί αυτό το σύστημα για τη βιομηχανία ενέργειας και για τη βιομηχανία γενικότερα. Από εκεί εξαιρούνται η κινητικότητα, οι μεταφορές δηλαδή και οι συγκοινωνίες. Επίσης εξαιρούνται τα κτίρια, η στέγαση, ε, η ηλεκτροδότηση και η θέρμανση και εξαιρείται και η γεωργία. Πιστεύω ότι για μια νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ένα νέο Κοινοβούλιο θα ήταν ενδιαφέρον να συζητήσετε μήπως το σύστημα εμπορίας ρήπων ε, να συμπεριλαμβάνει και τις εκπομπές ε, των μεταφορών αλλά και των κτηρίων για την ψήξη, για τη θέρμανση, για την ηλεκτροδότηση. Υπάρχουν ήδη κάποιες προσπάθειες σε κάποια κράτη-μέλη αλλά και πάλι στην εσωτερική αγορά για να έχει νόημα κάτι θα πρέπει να γίνεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Από εκεί θα έρθουν οι λύσεις. Τώρα, ε, ποια είναι τα μέσα που θα μπορούσε να σας προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο συνάδελφος Φρανς Τίμερμανς στη νέα Επιτροπή Φόντερ Λάιεν θα έχει την ηγεσία αυτού του χαρτοφυλακίου. Γι' αυτό είμαι κάπως επιφυλακτικός σήμερα, γιατί αρμόδιος για το Green Deal είναι ο κύριος Τίμερμανς. Στι πρώτε 100 ημέρε από την ανάληψη των καθηκόντων τη Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έρθει να σα τα παρουσιάσει αυτά και σε εσά και στο Συμβούλιο και στην κοινή γνώμη με ε, κάποιε αξιολογήσει και εκτιμήσει. Πάντω είναι γεγονό και είναι σαφέ ότι ε, ποντάρουμε πρώτα στην τεχνολογία. Σύγχρονη τεχνολογία, σύγχρονες τεχνολογίες που επιταχύνουν την ενεργειακή απόδοση, που σε βοηθούν πάρα πολύ. Το πρόγραμμα Horizon Ευρώπη είναι πάρα πολύ αποφασιστικό προς την κατεύθυνση αυτή, το ερευνητικό. Δεύτερον, ποντάρουμε ε, στο γεγονός ότι στο μέλλον θα συνεχιστεί το σύστημα ETS και θα αυξηθεί και η τιμή ε, ανά ανάλογα με τις νέες ποσότητες. Εδώ το Κοινοβούλιο ε, πρωταγωνιστεί στις συζητήσεις και θα συνιστούσα να ε, το ξανακάνετε. Τρίτον, έχουμε ένα στόχο μείωση 40% με τα μέτρα που είχαν αποφασιστεί στο ακόμα παλιό κοινοβούλιο, το πακέτο για την καθαρή ενέργεια, το πακέτο για την κινητικότητα, μπορούμε σύμφωνα με τους δικούς μας υπολογισμούς να φτάσουμε στο μείον 40% μέχρι το 2030 και μάλιστα 45%. Τώρα γίνεται η συζήτηση για 50% ή περισσότερο ακόμα. Εδώ χρειάζονται μελέντες αντικτύπου για να δούμε τι θα γίνει με τα πακέτα του περασμένου κοινοβουλίου, αυτές τις νομοθετικές δέσμε. αν χρειάζεται συνέχιση, συμπλήρωση ή και αναθεώρηση ακόμα. Πρόκειται επίση για εμπορικές συμφωνίες. Η Ευρώπη εκπέμπει παγκοσμίω μόλις το 9% των αερίων του θερμοκηπίου. Οπότε, μια εμπορική συμφωνία με άλλες χώρες, με άλλους εταίρους, και μια κοινή μείωση των εκπομπών έχει πάλι πάρα πολύ νόημα. Και ποτέ δεν ήταν αυτό πιο επίκαιρο. Σιγκαπούρη, Νέα Ζηλανδία, Μερκοσούρ, Μεξικό, μια σειρά χώρες είναι αυτές με τις οποίες διαπραγματευόμαστε ε, και συνάπτουμε συμφωνίες. Και μπορεί και αυτό το θέμα να αποτελέσει τμήμα των εμπορικών συμφωνιών. Θα πρέπει βέβαια να εξεταστεί ε, και για εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση εάν ε, ε, είναι θεμητός ο ανταγωνισμός αν αποφεύγεται η διαρροή του διοξιδίου του άνθρακα. Να δούμε μήπως χρειαστεί ένα τέλος διοξιδίου του άνθρακα. Η κυρία Φόντερ Λάιεν το είπε και στο κοινοβούλιο σας ότι αξίζει να εξεταστεί κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να εξεταστεί εάν συνάδει με τους κανόνες του ΠΟΕ, τι γίνεται με τον ανταγωνισμό και ενδεχομένως να είμαστε και πρόθυμοι να δεχτούμε εμπορικέ διενέξεις μέχρι και εμπορικού πολέμους. Γιατί δεν ξέρουμε πώς το βλέπει η Ουάσιγκτον ή κάποιοι άλλοι εταίροι. Ε, εκεί υπάρχει ένα πολιτικό κόστος που θα πρέπει να σταθμιστεί. Το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο που είναι υπό την αιγίδα της Προεδρεύουσας του Συμβουλίου, βρίσκεται σιγά σιγά στην τελική ευθεία το 25% όλων των επενδύσεων, όλων των δαπανών ε, έχουν ε, σχέση με το κλίμα. Από 160 δις ετησίως δηλαδή, ε, είναι 40%. Δεν είναι ευκαταφρόνητο ποσό. Σε ένα πρόγραμμα 40%, σε άλλο 60%, σε κάποιο άλλο 0%, γιατί μπορεί να μην έχει σχέση με την προστασία του κλίματος και του περιβάλλοντος εντός του δημοσιονομικού πλαισίου ε, ενδεχομένως να δημιουργηθεί ένα ταμείο δίκαιης μετάβασης. Υπάρχουν 41 περιφέρειες σε 12 κράτη-μέλη που είναι ανθρακοπαραγωγές και χρειάζεται να γίνουν μεταρρυθμίσεις, να ε, ε, προχωρήσουν. Σιγά-σιγά ε, να ε, φύγουμε από το θερμοελεκτρικό εργοστάσιο και το υδροελεκτρικό εργοστάσιο. Μάλλον για την παραγωγή ε, ρεύματος και θέρμανσης. Αλλά αυτά όλα θα πρέπει να γίνουν με δίκαιο τρόπο, με κοινωνική δικαιοσύνη και σεβασμό. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπονεί ε, σχετικά έγραφα αυτό τον καιρό για το πώς θα μπορεί να έχει ένα ταμείο δίκαιης μετάβασης, πώς θα υιοθετηθεί και ποιοι θα είναι οι όροι για να αντλούνται πόροι από αυτό το ταμείο. Και εδώ θα είναι ευπρόσδεκτη η δική σας συνεισφορά τις επόμενες εβδομάδες. Την εκτιμούμε τα μάλα. EU Invest, επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τράπεζες, διαθροτικές, θα είναι σίγουρα ένα τμήμα των εργαλείων και των μέσων του νέου πράσινου deal. Πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει δημόσιου πόρους, ευρωπαϊκούς, κρατικούς, περιφερειακούς και να τους συνδυάσει με ιδιωτικούς με την καλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα. Με δύο λόγια, δεν τελειώνει εδώ αυτή η υπόθεση. Τώρα αρχίζει. Η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή Φοντερ Λάιεν και ο Φρανς Τίμερμας θα είναι οι συγκεκριμένοι συνομιλητές σας για να συνεχιστεί η προσπάθεια της προηγούμενης Επιτροπής και του προηγούμενου Κοινοβουλίου ε, κρατώντας την κατεύθυνση αλλά ενδεχομένως επιταχύνοντας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Τώρα, από τις πολιτικές ομάδες και εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, για δύο λεπτά το λόγο έχει η κυρία Ντελάνγκε. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είναι σαφέ ότι η αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών είναι από τι μείζονε προκλήσει των καιρών μα. και πολύ σωστά αναφέρθηκε ότι είναι και ύψιστη προτεραιότητα τη Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ω Χριστιανοδημοκράτησα, πιστεύω ότι ο πλανήτη δεν είναι ιδιοκτησία μα. Τον κρατούμε και το φροντίζουμε για τι επερχόμενε γενιέ και έχουμε ηθικό καθήκον να τον φροντίσουμε. Στη συζήτηση αυτή είμαι βέβαιη ότι κάποιοι θα ε, αδιαφορήσουν, θα περιφρονήσουν τις επόμενες γενιές ε, λέγοντας ότι δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή, δεν είναι πρόβλημα και θα αρνηθούν να λάβουν μέτρα. Υπάρχουν όμως και άλλοι που θα σας πούν τι θα έπρεπε να κάνουμε ε, και τι να αποφύγουμε. Θα πρέπει να θερμομονώσουμε τα σπίτια μας, να αγοράσουμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τέσλα, ενώ άλλοι δεν έχουν να φάνε στο τέλος του μήνα. Υπάρχει όμως και τρίτος δρόμος, αυτό, αυτή είναι η δική μας άποψη, που μπορεί να μετριάσει και να αντιμετωπίσει κλιματικές αλλαγές, αλλά χωρίς να επιβαρύνει τους ε, απόρους, εκείνους που δεν μπορούν να αναλάβουν αυτό το βάρος και να βοηθήσουμε τον κόσμο. Γι' αυτό μιλούμε για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης κατά τη γνώμη του ΕΛΚ, δεν θα πρέπει να έχουμε μόνο μια Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και κλιματικού στόχου, αλλά και μια ισχυρή βιομηχανική στρατηγική, ώστε να φροντίσουμε να έχουμε την καθαρότερη και την πιο καινοτόμα βιομηχανία που θα διαφυλάσει θέσει απασχόληση για τι μελλοντικέ γενιέ που θα τι χρειαστούν. Και αν ε, συνάδελφοι που μιλούν για αηφορία και βιωσιμότητα ε, ναι, όντω, η βιωσιμότητα έχει και περιβαλλοντικό χαρακτήρα, αντιμετωπίζει την κλιματική αλλαγή, αλλά θα πρέπει να μιλήσουμε και για οικονομική και και κοινωνική βιωσιμότητα. Χρειαζόμαστε μια ισχυρή βιομηχανία για να υλοποιήσουμε τους στόχους μας κατά της κλιματικής αλλαγής. Οπότε αν ε, οι συνάδελφοι είναι πρόθυμοι να επεξεργαστούμε και τις τρεις αυτές πτυχές, ε, το ΕΛΚ θα είναι σημαντικός σύμμαχος και εταίρος στη διαδικασία αυτή. Εκ μέρους των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και για δύο λεπτά το λόγο έχει η κυρία Φριτσό. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ ε, τρέφω μεγάλο σεβασμό προς τη Διακυβερνητική Επιτροπή των Ηνωμένων Αθηνών για την Κλιματική Αλλαγή. Θεωρώ ότι υπάρχει ακόμη δυνατότητα να αντιστρέψουμε τις τάσεις ε, και να υλοποιήσουμε τους στόχους της Συμφωνίας των Παρισίων. Ω σοσιαλίστρια είναι σημαντικό ότι η Ευρώπη θα πρέπει να δείξει το καλό παράδειγμα, να γίνουμε υπόδειγμα και να έχουμε μια κοινωνία που θα προστατεύει και το κλίμα. Θα πρέπει φυσικά να μειώσουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στα πλαίσια της ενεργειακής μας πολιτικής. Θα πρέπει να στραφούμε προς πιο φιλοπεριβαλλοντικές και καθαρές πηγές ενέργειας. Θα πρέπει να περιορίσουμε τις εκπομπές από τις μεταφορές και τις ρηπογόνες εκπομπές. Είναι προφανές ότι θα πρέπει να έχουμε πιο δραστική και πιο γρήγορη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από ό,τι μέχρι σήμερα, για να τηρήσουμε τη Συμφωνία των Παρισιών. Για να γίνουν όλα αυτά όμως θα πρέπει να δείξουμε τον πολιτικό δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε. Εμείς σοσιαλιστές είμαστε έτοιμοι. Είναι προφανές ότι θέλουμε μια οικολογική κοινωνία που δεν θα αμελεί όμως τον άνθρωπο. Είμαστε πεπισμένοι ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε με συνεργασία και να επιτύχουμε ταυτόχρονα τη μείωση των εκπομπών και την αύξηση τη οικονομική μα ανάπτυξη. Έτσι μπορούμε να δημιουργήσουμε νέε θέσει απασχόληση. Έτσι θα μπορέσουμε να αλλάξουμε την αγορά εργασία. Δική μα ευθύνη είναι να βοηθήσουμε τους πολίτες να αναπτύξουν νέες δεξιότητες ώστε να αντιμετωπίσουν αυτές τις αλλαγές. Είναι σημαντικό επίσης να αντιληφθούμε ότι αυτός ο στόχος ε, είναι αξιοσημείωτος. Ε, είμαι Σουηδέζα η σοσιαλιστική μας κυβέρνηση είναι υπέρ των κλιματικών προσπαθειών και υπέρ των επενδύσεων για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Πιστεύω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε όλοι μαζί και να αποδείξουμε στην Κρέτα και σε όλους τους νέους ότι είμαστε πρόθυμοι να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή. Εκ μέρους του Ρήνιο και για δύο λεπτά το λόγο έχει η κυρία Ροντρίγκε Ράμος. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι. Η ομάδα μου γνωρίζει ότι κανεί δεν θα πρέπει να παραμείνει στο περιθώριο. Κανένα θεσμικό όργανο, κανένα νομοθέτη, καμία κυβέρνηση δεν θα πρέπει να μείνει στο περιθώριο αυτή τη καταστροφή που προκαλεί η κλιματική αλλαγή και που ήδη προκαλεί μεγάλη οδύνη. Έχουμε ελάχιστη χρόνο για να ελέγξουμε αυτή την υπερθέρμανση του πλανήτη και αν θέλουμε να την αναχαιτήσουμε θα πρέπει να δράσουμε αμέσως με πολύ συγκεκριμένα εκτεταμένα μέτρα πρωτοφανή για τα μέχρι τώρα δεδομένα. 93% των Ευρωπαίων πολιτών θεωρούν ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το πρόβλημα, αλλά κυρίως οι νέοι, τα παιδιά μας θεωρούν ότι το πρόβλημα είναι και κατεπήγον, γιατί διανύουμε μια πραγματική κλιματική κρίση. Υπάρχει έκτακτη ανάγκη και γι' αυτό οι νέοι μας κάθε, μέρα, κάθε Παρασκευή κατεβαίνουν στους δρόμους για να απαιτήσουν δράση από εμά. Έχουμε ένα πεπερασμένο πλανήτη και έχουμε υπερβολικά μεγάλο αριθμό αποβλήτων και καταναλώνουμε πολλούς πόρους. Σε μερικούς παραγωγικούς τομείς ε, σπαταλούμε το 98% της παραγωγής μας. Πώς λοιπόν θα καταφέρουμε να εξορθολογήσουμε την παραγωγή μας και την κατανάλωσή μας. Θέλουμε ένα σύστημα κυκλικής οικονομίας. Θα πρέπει να περάσουμε από την ανακύκλωση στην πρόληψη, να ασθενιστούμε τη βιοοικονομία, ώστε ό,τι χρησιμοποιούμε και όλοι μας οι φυσικοί πόροι να τη χάνουν προστασίας και συντήρησης από όλα τα συστήματα παραγωγής. Θα πρέπει διαφορετικά να σχεδιάσουμε τις πόλεις μας, να είναι πιο πράσινες, γιατί το 70% των πολιτών μένουν στις πόλεις. Επίσης, θα πρέπει να απαλλαγούμε από τις εκπομπές άνθρακα να έχουμε μηδενικέ εκπομπέ άνθρακα στην οικονομία μα. Και αυτό θα πρέπει να γίνει οριζόντια σε όλου του τομεί. Γιατί έχουμε ένα πρόβλημα. Δεν έχουμε μια δεσμευτική παγκόσμια διακυβέρνηση. Οι συμφωνίε που συνάπτουμε είναι προαιρετικέ. Γι' αυτό και είναι σημαντική η Σύνοδο Κορυφή των Ηνωμένων Εθνών. Μα λένε τα Ηνωμένα Έθνη. Θέλετε περισσότερε συμφωνίε, πιο, πιο ε, άμεσες και πιο αποφασιστικέ. Εμεί δίνουμε ένα καλό χάρτη, μια καλή πηξίδα για το θέμα αυτό με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Θα πρέπει όμω να έχουμε επίγνωση ότι χωρί τη συμφωνία και τη δέσμευση όλων των κρατών μέλων δεν θα έχουμε αναμενόμενα θετικά αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Εκ μέρου των Πρασίνων τώρα, ο κ. Έκχαουτ για δύο λεπτά. Uh, Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ που προβλέψατε το σημείο αυτό στην ημερήσια διάταξη υπό τον τίτλο «Κλιματική και οικολογική κατεπήγουσα ανάγκη». Γιατί πρέπει να είμαστε πραγματικά εδώ ειλικρινεί. Όταν ακούω να μιλάτε δεν αισθάνομαι ότι έχετε αντιληφθεί ότι έχουμε κάτι το κατεπήγον εδώ να αντιμετωπίσουμε προς το κλίμα. Ε, η Επιτροπή μιλάει για στόχους που θα εφαρμοστούν και θα επιδιωχθούν οι οποίοι αποφασίστηκαν πριν από πέντε χρόνια επιστήμη έχει προχωρήσει. Διαβάστε όλες τις επιστημονικές μελέτες που εκδίδονται καθημερινά Κοιτάξτε που λένε, πώς λένε ότι αντιμετωπίζουμε μια κατεπίγουσα ανάγκη. Μιλάμε για το μέλλον μας, αλλά έχουμε και ευκαιρίες. Ευκαιρίες η Ευρωπαϊκή Ήπειρος να αλλάξει την οικονομία της, να βασιστούμε στην κλιματική μενιβωτερότητα, αλλά να δημιουργήσουμε και νέες θέσεις εργασίας. Υπάρχουν ένα σωρό μελέτες και ακόμα το Συμβούλιο πασχίζει για να συμφωνήσει για την κλιματική ουδετερότητα. Ίσως τώρα το Δεκέμβριο, ε, μέσα σε ένα χρόνο θα τα καταφέρει και μέχρι το χρόνο κάτι να έχει ξεκινήσει. Μα με τον ίδιο στόχο που συμφωνήσαμε πριν από πέντε χρόνια θα προχωράμε. Αυτό δεν είναι αναγνώριση τη κατεπίγουσα ανάγκη, αυτό που ζητάνε οι πολίτε. Πρέπει να γίνουν περισσότερα το κατεπήγον πρέπει να το αντιληφθούμε με σαφήνεια και όχι με τα λόγια και τις κουβέντες εδώ αλλά με δράση από το Συμβούλιο, την Επιτροπή και από το ίδιο το σώμα μας. Ωραία να ακούμε όλες αυτές τις ομιλίες που έχουμε εδώ στην Ολομέλεια αλλά όταν μιλάμε για πολιτική το σώμα μας δεν κάνει τίποτα. Τη στιγμή αυτή που συζητάμε για την γεωργία, τη μεταρρύθμιση της αγροτικής πολιτικής, ο τομέας της γεωργίας είναι σημαντικός και μπορεί να προσφέρει για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Ζητώ λοιπόν από τους συναδέλφους να εγκρίνουν μέτρα που θα να μα επιτρέψουν να πετύχουμε αποτελέσματα. Όχι μόνο στα λόγια εδώ, στι ομιλίε μα εδώ πέρα, αλλά η γεωργία πραγματικά να πάρει πράσινη μορφή και όχι απλώ να επιδοτούνται για άλλη μια φορά οι μεγάλε εκμεταλλεύσει. Και το τελευταίο για το εμπόριο, να βεβαιωθούμε ότι οι εμπορικέ μα συμφωνίε πραγματικά συνάδουν με του κλιματικού μα στόχου. Σταματήστε με αυτά τα κεφάλαια περί αηφορία να γίνουν δεσμευτικά, ώστε διεθνώ να πιέσουμε για τι προτεραιότητέ μα με την κατεπίγουσα πραγματικά ανάγκη που αξίζει αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε εκ μέρους της ID η κυρία Σαρντόνε για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Οι σοσιαλιστές πρότειναν και πέτυχαν το βασικό θέμα της Ολομέλειας αυτής να είναι η κλιματική και οικολογική κατεπήγουσα ανάγκη, το κατεπήγον. Όμως ε, η αριστερά κάποτε ασχολείται με τους αδύναμους, τους εργαζομένους, το λαό. Τι έχει αλλάξει. Εδώ πραγματικά ήλπιζα ότι η αριστερά θα πρόβλεπε μια συζήτηση για τα κοινωνικά δικαιώματα, τους μισθούς, για τις κοινωνικές εισφορές. Μάλλον η φτωχή δεν είναι πλέον της μόδας. Η Γκρέτα έχει συμπαρασύρει μαζί τη όλου αυτού που τώρα διαδηλώνουν για να, ως μαθητές να, κάνουν κοπάνα από το σχολείο. Εδώ λοιπόν έχει φέρει αυτό το θέμα στην πρώτη γραμμή για όλη την Ευρώπη. Ολόκληρη η ήπειρο, ε, όπω λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρέπει να εφαρμόσει προγράμματα τα οποία είναι ανέφικτα, με μη ρεαλιστικούς στόχους, ε, προγράμματα τα οποία είναι περιτά και πολλέ φορέ με λανθασμένους στόχους. Η παραγωγή και η πραγματικότητά τη είναι σημαντική και το κόστο που θα πληρώσουν οι καταναλωτέ με το πλέον σημαντικό. Πώ θα προσπιστούμε το περιβάλλον. Και εμεί θέλουμε να το προστατεύσουμε. Αλλά όχι με πολιτικέ των συνθημάτων που απλώ βασίζονται σε φόρου και περιβαλλοντικέ φιλοδοξίε. Καλύτερα να βάλουμε τι σωστέ προτεραιότητε και να αφήσουμε τα κατεπήγοντα. Ευχαριστούμε εκ μέρου των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών για 1,5 λεπτό ο κύριος Βόντρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εμείς συντηρητικοί είμαστε και θεωρούμε φυσικά ότι θα πρέπει να μεταβιβάσουμε το περιβάλλον στα παιδιά μας, όχι σε χειρότερη κατάσταση, αλλά σε καλύτερη από εκείνη που εμείς το κληρονομήσαμε. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να πω ότι το πράσινο deal θα είναι πανάκριβο και μπορεί ε, να πλήξει τους ανθρώπους χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος σε διάφορες χώρες αναδυόμενες και μπορεί να αποδειχθεί και άχρηστο εγχείρημα εάν η Κίνα, οι Ηνωμένε Πολιτείε και λοιποί δεν μας ακολουθήσουν. Για το λόγο αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξει σωστή αξιολόγηση και εκτίμηση αντικτύπου των δραστηριοτήτων μας, δεν χωράει καμία αμφιβολία, να έχουμε ένα πρόγραμμα για το τι θα κάνουμε με τα πιο ευάλωτα κράτη-μέλη και τους ανθρώπους χαμηλού εισοδήματος στις κοινωνίες μας, και επίσης κάτι άλλο που δεν είναι λιγότερο σημαντικό, δεν έχει κανένα νόημα τώρα να επιταχύνουμε τις δεσμεύσεις μας εάν δεν δεσμευθούν σαφώς οι άλλοι. Που δεν υπάρχει. Υπάρχει μια τσεχική παροιμία που λέει ότι ο δρόμος προς την κόλαση είναι στρωμένος με καλές προθέσεις. Και θυμάμαι ότι ο πρόεδρος Μακχόν ε, είχε εφαρμόσει πάρα πολύ λίγα μέτρα σε σχέση με αυτά που εμείς τώρα εξαγγέλουμε και του βγήκαν αμέσω τα κίτρινα γυλαίκα στο δρόμο. Ε, ε, λοιπόν, είναι πολύ ε, επικίνδυνο να δούμε σκηνές της περσινής χρονιάς και φέτος. Εξ ονόματος της ΓΟΕ, για ένα λεπτό, η κυρία Ματίας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Έτιγκερ, μπορεί να εκπλαγείτε, αλλά πραγματικά είναι απογοητευτικό. Αισθανόμαστε πραγματικά φρούστρα κάθε φορά που σα ακούμε να μιλάμε για τα κλιματικά και το περιβάλλον. Ε, το κατεπήγον θέμα θα τα αντιμετωπίσουμε με παλιές λύσεις που δεν λειτουργήσανε και τις ξαναδοκιμάζουμε εδώ. Θέλουμε να μας πείτε ποιες είναι οι προτεραιότητες και εσείς μας μιλάτε για την ε, αγορά, μιλάμε για εμπορικές ποσοστώσεις, μιλάμε για όλα αυτά που μας οδήγησαν σε αυτή την καταστροφή και ακόμα δεν έχουμε βρει μια λύση. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το κατεπήγον των κλιματικών αλλαγών, κύριε Έτιγκερ, με μέτρα πράσινη οικονομία που δεν αλλάζουν σε τίποτα το σύστημα, που δεν αλλάζουν τι δημόσιε επενδύσει, που δεν προβλέπουν την ενεργειακή διαφοροποίηση και δεν προβλέπουν καμία ε, περιβαλλοντική δικαιοσύνη, ή κοινωνική δικαιοσύνη. Πρέπει να ακούσουμε τον κόσμο που βρίσκεται στου δρόμου. γιατί είναι σημαντικό τώρα να τους αφουγκραστούμε. Ιδάλω δεν θα έχουμε κανένα πλανήτη για να μπορέσουν να ζήσουν οι μελλοντικέ γενιέ αν τώρα δεν κάνουμε κάτι. Κύριε Έτιγκερ, δεν φτάνει να παίζουμε με τι πράσινε συμφωνίε εάν δεν έχει καμία ε, ρεαλιστική πορεία για να ακολουθήσει αυτό το Green Deal. Ευχαριστούμε από και γραμμέ για 1,5 λεπτό η κυρία Εύη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ε, συμφωνώ με όσα είπαν ε, οι συνάδελφος Ματίας ο κύριο Σέικχαουτ. Πραγματικά είναι τελείω αναχρονιστικό να συζητάμε τώρα για ένα σύστημα εμπορικό των εκπομπών που δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα. Είναι σαν να πηγαίνουμε πίσω στο παρελθόν και να μην αντιμετωπίζουμε το κατεπήγον που έχουμε μπροστά μα. Για να αντιμετωπίσουμε όμω αυτό το κατεπήγον θα πρέπει να σκεφτούμε και θέλω να το θέσω επιτάπητο σε ένα ακόμα ζήτημα, το έδαφο. Διότι η αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών δεν μπορεί να με λαμβάνει υπόψη την προστασία του εδάφου, τη γη. Εδώ χρειάστηκαν 2000, χρειάζονται 2.000 χρόνια για να δημιουργήσουμε με δύο ε, εκατοστά εγών εδάφου και αυτό μπορεί μια πλημμύρα να το συμπαρασύρει. Όπω έγινε πρόσφατα πριν από λίγε μέρε στη Λομπαρδία στη Λιγουρία. Εδώ λοιπόν πρέπει η Ευρώπη να σκεφτεί τις το ότι κάθε χρόνο έχουμε το ισοδύναμο 270 γηπέδων ποδοσφαίρου που μολύνονται ε, ο έδαφος κάθε χρόνο, κάθε μέρα. Θα πρέπει λοιπόν αυτό να το σκεφτούμε. 24% του εδάφους το χάνουμε, αλλά δεν είναι μόνο το πρόβλημα του εδάφους στην Ιταλία, είναι και στην Ισπανία, στη Γαλλία και σε όλες τις υπόλοιπε χώρες που ζουν τις ίδιες συνθήκες. Ξέρω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ξεκινήσει μια στρατηγική για την βιοπικιλότητα. Θα πρέπει να λάβει υπόψη της και την προστασία του εδάφους, διότι είναι το 1 τέταρτο της βιοπικιλότητας ε, αυτό και θα πρέπει να προβλέψουμε ένα στόχο ουδετερότητας για την προστασία του εδάφου μέχρι το 2030. Διότι χωρί ακριβώ αυτή την προστασία δεν μπορούμε να αναχαιτήσουμε τι κλιματικέ αλλαγέ και για να το κάνουμε χρειαζόμαστε μια πολιτική σφαιρική η οποία να αντιμετωπίσει την εντατική κτηνοτροφία, την μονοκαλλιέργεια και τη χρήση λοιπασμάτων χωρί έλεγχο. Ευχαριστώ. For a minute and half. Για 1,5 λεπτό η κυρία Βάις. Αλλαγή του ομιλητή. Ευχαριστώ. Συνάδελφοι, ευτυχώς που συζητάμε το κλίμα και την προστασία του περιβάλλοντος σήμερα. Είναι ένα σημείο κρίσιμο στη φάση της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Πρέπει λοιπόν να θέσουμε μεταξύ μας τις σωστές ερωτήσεις, να βρούμε τις σωστές απαντήσεις και να συζητήσουμε για να καταρτήσουμε τη σωστή ε, γραμμή δράσης. Εδώ πρέπει να σκεφτούμε πώς θα προστατεύσουμε το περιβάλλον χωρίς να χάσουμε θέσεις εργασίας και κάτι τέτοιο είναι εφικτό. Πρέπει και οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε τις περιβαλλοντικές προκλήσεις ε, και να δούμε τις ε, δυνατότητες δημιουργίας θέσεων εργασίων, ε, Πρέπει να εκμεταλλευτούμε όλες τις δυνατότητες και για την οικονομία και μην ξεχάσουμε τις 9.000, τις 900.000 θέσεις επιχειρήσεις που σχετίζονται με αυτό το τομέα και είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας. Η ε, ευφυής χρήση όλων αυτών των μέσων θα μας επιτρέψει να αποφύγουμε την περαιτέρω μείωση θέσεων εργασίας και να, να εξοπλίσουμε όλες τις ευκαιρίες. Είναι λίγο προφανής αυτή η λογική, την βλέπει και το ΕΛΚ και ελπίζουμε να καθοδηγήσει και την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία πιστεύοντας στο ελεύθερο εμπόριο και την ε, προώθηση των ε, ελεύθερων συναλλαγών μπορεί να προωθήσει και την προστασία του περιβάλλοντος ταυτόχρονα σε όλο τον πλανήτη. Ευχαριστώ. για δύο λεπτά κυρία Γκούτελαντ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πραγματικά θα ήθελα να δράσουμε άμεσα σαν να καίγεται το σπίτι μας. Αυτά είναι τα λόγια της Γκρέτα Τούμπερκ. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Το σπίτι μας έχει πάρει φωτιά. Δεν μπορούμε να μένουμε με τα χέρια σταυρωμένα. Βλέπουμε εκατοντάδες επιστημονικές μελέτες που επιβεβαιώνουν το ίδιο ακριβώς πράγμα. Ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο κόσμος ολόκληρος θα πρέπει να την αντιμετωπίσει. Είναι εύκολο να ε, νιώθουμε ανήμποροι, να υποκύψουμε ε, στην ε, απελπισία. Αλλά μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα μέλλον με περισσότερη ευημερία, οικονομική ανάπτυξη και θέσει απασχόληση στην Ευρώπη. Για να το επιτύχουμε όμω, θα πρέπει να γίνουμε πρωτοπόροι, να πρωτοστατήσουμε και να δείξουμε το σωστό δρόμο και να υιοθετήσουμε τα σωστά μέτρα, γιατί έχουμε συγκεκριμένες ευθύνες και καθήκον. Επίσης, θα πρέπει να επενδύσουμε στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Αν δεν προασπίσουμε την καινοτομία, αν δεν δημιουργήσουμε φιλοπεριβαλλοντικές θέσεις εργασίας που χρειάζονται για να μείνουμε ανταγωνιστικοί, και να βρεθούμε στην αιχμή τη αλλαγή, δεν πρόκειται να τα καταφέρουμε. Για μας, του Σοσιαλιστέ και δημοκράτε, τα πράγματα είναι φω φανάρι. Έχουμε ευκαιρία και θα πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι. Γι' αυτό απαιτούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερε φιλοδοξίε. Θα πρέπει να μειώσουμε τουλάχιστον κατά 55% τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα μέχρι το 2030. Θα πρέπει να σταματήσουμε τι επιδοτήσει που δίνονται ακόμη σε τομείς που χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα. Γιατί τέτοιου είδους επιδοτήσεις αντιβαίνουν στις κλιματικές μας δράσεις που είναι απαραίτητες. Ακόμη και σήμερα έχουμε κάποιους τομείς που περνούν απαρατήρητοι. Θα πρέπει όμως να τους θέσουμε στο στόχαστρο και να θέσουμε και για αυτούς τους τομείς συγκεκριμένους στόχους, ποσοτικοποιημένους, για την αεροπορία, για παράδειγμα, θα πρέπει να είμαστε πιο απαιτητικοί. Είναι σημαντικό για το κλίμα. Έχουμε μια ευκαιρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση να δράσουμε και να γίνουμε πρωτοπόροι. Δεν πρέπει να τη χάσουμε. Ευχαριστώ, κυρία Σαμπό. Σα ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ω προ την κλιματική έκτακτη ανάγκη, έχω στο μυαλό μου την ίδια εικόνα συνεχώ. Είμαστε σαν το ναυτικό που βλέπει την καταιγίδα να καταφθάνει, αλλά δεν μειώνει την ιστιοφορία του περνάνε μήνες και χρόνια ολόκληρα, αλλά εμείς εκεί δεν πρόκειται να μειώσουμε τα, τα πανιά μας, ούτε να υιοθετήσουμε τη σωστή ταχύτητα. Παρ' όλα αυτά, έχουμε την ευαισθητοποίηση να γενικεύεται. Πολλές χώρες να έχουν βάλει ως στόχος του, ως στόχος του στην ουδετερότητα του άνθρακα για το 2050. Και αυτή είναι η προτεραιότητα και της Μελλοντικής Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχουν όμω λύσει. Αν μειώσουμε κατά δύο κόμβου τη ταχύτητα των πλοίων, θα έχουμε κατά 20% εξοικονόμηση των εκπομπών τη ναυσιπλοεία. Επίση, μπορούμε να μειώσουμε τη χρήση των κλιματιστικών, γιατί τα κτίρια και τα δημόσια κυρίω κτίρια είναι, έχουν υπερβολική θέρμανση, υπερβολική ψήξη με την υπερβολική χρήση των κλιματιστικών. Θα πρέπει λοιπόν να αναλάβουμε αυτά τα μέτρα για να συγκρατήσουμε την αύξηση της θερμοκρασία του πλανήτη στον 1,5 βαθμό. Κάθε μισός βαθμός μετράει. Αυτό μας ε, υπενθύμησαν και στη Νέα Υόρκη. Θα πρέπει λοιπόν εν ώψη τη επόμενη διάσκεψη κορυφή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση να πρωτοστατήσουν στην προσπάθεια για, την, για τον έλεγχο των κλιματικών αλλαγών. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ζαντό. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε το κατεπήγον που πρέπει να συζητήσουμε σε αυτή τη Σύνοδο Ολομέλεια δεν είναι το κατεπήγον των επιστημονικών πορισμάτων. Το γνωρίζουμε όλοι. Είναι το κατεπήγον τη δράση που απαιτείται. Δράση και ξαναδράση και πάλι δράση. Εδώ λοιπόν άκουσα τον Επίτροπο Έτιγκεν να μα κάνει τον απολογισμό τη απερχόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να είναι αυτό το φύλλο πορεία τη κατεπήγουσα δράση που χρειαζόμαστε για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Δεν ε, ε είμαστε στη σωστή τροχιά για την ε, Συμφωνία των Παρισίων. Οι προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη δική σα Επιτροπή για την κοινή αγροτική πολιτική ενισχύουν τι αρνητικέ επιπτώσει τον εκπομπών του θερμοκηπίου και την απώλεια τη βιοπικιλότητα. Κάνουμε ακριβώ το αντίστροφο. Υποστηρίζεται συμφωνίε ελεύθερων συναλλαγών που είναι κλιματοκτόνε και πραγματικά ε, οδηγείται στην εξουδετέρωση, την, ε, τον αφανισμό τη βιοπικιλότητα. Χρησιμοποιείται εκατομμύρια, δισεκατομμύρια ευρώ για τον ε, διάσωση των τραπεζών. Να χρησιμοποιήσετε τα δισεκατομμύρια ευρώ για τη διάσωση του κλίματο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μπορούν να χρηματοδοτήσουν ένα ευρύ ε, πρόγραμμα επενδύσεων ε, που να δημιουργήσει και αγοριστική δύναμη και επενδύσει και να ενισχύσει του καταναλωτέ και να αντιμετωπίσουμε και τον Πούτιν και όλου του άλλου για το καλό τη Ευρώπη, για το καλό του κλίματο. Πρέπει να υπάρχει όμω πολιτική βούληση. Για ένα λεπτό η κυρία Γκριζέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Συμφωνούμε όλοι για να κηρύξουμε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το κλίμα. Λιγότερο συμφωνούμε ως προς τα μέτρα και την αποτελεσματικότητά τους. Για τα οικονομικά αυτού του πράσινου συμφώνου, πώς θα βρούμε ένα 3 εκατομμύριο ευρώ αυτή τη στιγμή που δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε ένα πράσινο ταμείο 10 φορές μικρότερο. Πώς θα φτάσουμε χωρίς να έχουμε περισσότερη Ευρώπη και περισσότερη φορολογία με πρόφαση την οικολογία. Η οικολογική προτεραιότητα πρώτα απ' όλα είναι να δούμε ε, πώς αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο ο παγκόσμιος πληθυσμός. Από την άλλη θα πρέπει να ξεφύγουμε από την παγκοσμιοποίηση για τις εμπορευματικές ροές και τις ανθρώπινες και να ξαναγυρίσει η τοπική παραγωγή, τοπική συνεργασία, κρατική συνεργασία με συγκεκριμένους στόχους ε, και καλή διάγνωση και έτσι μόνο θα μπορέσουμε να απαντήσουμε στις οικολογικές προκλήσεις. Για ένα λεπτό η κυρία Ζαλεύσκα. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επιτροπέ, κυρίες και κύριοι, κρίμα που είμαστε τόσο λίγοι στην αίθουσα. Τα παιδιά και οι νέοι που διαμαρτύρονται, αλλά και οι πολίτες που μας επέλεξαν, δεν περιμένουν από μας ημίμετρα ή απλώς διάπειρους λόγους. Περιμένουν απτά μέτρα, συγκεκριμένα σχέδια που επίσης θα περικοδοτούνται με, με τα απαραίτητα κονδύλια. Γι' αυτό προτείναμε και το Ταμείο Δίκαιη Μετάβαση. Από αυτό θα πρέπει να ξεκινήσουμε. Και τι έχουμε όμω, τίποτα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα λοιπόν οι Γάλλοι να συζητήσουν το θέμα αυτό με τον πρόεδρο Μακρόν και να ορίσουν τον επόμενο υποψήφιο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Γάλλο υποψήφιο επίτροπο, γιατί δεν έχουμε ακόμη επιτροπή. Θέλουμε συγκεκριμένο προπολογισμό και όχι απλώ συνθήματα και λόγια ωραία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όταν ρωτήσαμε τον Φραν Τίμερμαντ ε, τι μορφή θα έχει το περιβαλλοντικό νομοσχέδιο και πώς θα εξασφαλιστούν τα χρήματα για την προστασία του περιβάλλοντος, δεν απάντησε τίποτα ο κύριος Τίμερμανς, τίποτα συγκεκριμένο. Ελπίζω λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματικά θα εγγύψει με συγκεκριμένα μέτρα και προτάσεις στο θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος. Κυρία Χάζακαμ, για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όταν καίγεται το σπίτι σου, μετράει κάθε δευτερόλεπτο. Πώς είναι δυνατόν εδώ να συνεδριάζουμε χρόνια ολόκληρα για ασθενεί συμβιβασμού ενώ ο κόσμος μας καίγεται. Έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα. Και θα πρέπει να εξαγγείλουμε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη βιοπικιλότητα και για το κλίμα. Ένα εκατομμύριο ε, είδη απειλούνται με εξαφάνιση. Η κλιματική κρίση απειλεί δισεκατομμύρια ανθρώπου ζώα και φυτά σε όλα τα επίπεδα, σε όλα τα μέτωπα χρειάζεται δράση. Πώς είναι δυνατόν η Ευρώπη να δίνει δισεκατομμύρια ε, επιδοτήσεις ε, στη βιομηχανική κτηνοτροφία. Φλέγεται ο Αμαζόνιος για να έχει η Ευρώπη φτηνές ζωοτροφές και φτηνό κρέας. Η κτηνοτροφία παγκοσμίω ε, ευθύνεται για περισσότερα ε, αέρια του θερμοκηπίου από όλα τα αυτοκίνητα, ε, τρένα και καράβια και αεροπλάνα μαζεμένα. Πώς είναι δυνατόν ο κύριος Τίμερμανς να μην θέλει να μειωθεί ο αριθμός των ζώων που εκτρέφονται. Ε, πώς δεν καταλαβαίνουμε το κόστος κτηνοτροφίας. Μπορούμε να μειώσουμε το κόστος στο μισό αν τρώμε λιγότερο κρέας, λιγότερο ψάρι και λιγότερα γάλακτοκομικά και να περάσουμε στα φυτικά προϊόντα. Και δεν χρειάζεται αυτό χρόνια για να γίνει. Μπορούμε να αρχίσουμε κάθε δευτερόλεπτο. Και θα πρέπει η Ευρώπη αυτό να το ενθαρρύνει ε, ε, Σταματώντα τις επιδοτήσει για τα γαλακτοκομικά και το κρέας. Και κατά τα άλλα πιστεύω ότι θα πρέπει να καταργηθούν τελείως οι επιδοτήσει στη Γεωργία, στην Ευρώπη. Ευχαριστώ για 1,5 λεπτό. Ρόουλαντ, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όλες οι συζητήσεις για την κλιματική αλλαγή ε, μιλούν για την αποκάλυψη και τον Αρμαγεδόνα αν δεν αλλάξουμε ριζικά ε, το ενεργειακό μας και ε, τον τρόπο που ζούμε. Από το 1988 στο Τορόντο στη Σύνοδο που είπανε ότι θα είναι σαν πυρηνική καταστροφή. 1,5 με 4,5 βαθμούς Κελσίου λέει θα έχει αυξηθεί ε, μέχρι το 2030 η θερμοκρασία. Ε, τώρα είμαστε στο 0,25 μόλις ε, στο μισό του διαστήματος αυτού. στη δεκαετία του 70 μα είπαν οι επιστήμονες ότι μπαίνουμε σε εποχή των παγετώνων και θέλανε να ρίξουν στάχτη ε, στους πόλους, ε, ε, στους πάγους. Και τότε έξω πέσανε και τώρα έξω πέφτουνε. Δεν είναι δυνατό να μιλάμε για φαινόμενα ανθρωπογενή. Είναι και αστρονομικά τα φαινόμενα αυτά και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να μην αλλάξουμε τακτική. Κοιτάξτε να δείτε, η εγκατάλειψη του άνθρακα σημαίνει εγκατάλειψη ε, του πολιτισμού. Είναι ε, μονομερής αφοπλισμός. Καταθέτουμε τα όπλα και με επιδοτήσεις ε, των φορολογουμένων ε, θέλετε να επιδοτήσετε τους παραγωγούς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αυτοί οι καιροί ε, θα μείνουν στην ιστορία ως η πιο δαπανηρή ανοησία και φαύλος κύκλος που έκανε ποτέ κυβέρνηση σε αυτόν τον κόσμο. Για 1,5 λεπτό τώρα κυρία Μαγκίνες. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι ξεχνούμε τι συμβαίνει στον πραγματικό κόσμο. Για παράδειγμα, σήμερα η τοπική μου αυτοδιοίκηση έχει ένα ε, σεμινάριο για την κλιματική αλλαγή για τους ε, ε, υπαλλήλους του. Επίσης, η γειτονική επαρχία έχει πρωτοβουλίες που βοηθούν τις ευάλωτες κοινότητες, ευάλωτες οικογένειες να ανακαινήσουν τα σπίτια τους με ε, καλύτερη ε, θερμομόνωση. Ας μην, είμαστε, ας μην αψηφούμε λοιπόν αυτοί ε, τους υπόλοιπους, τις καταστάσεις. Επίσης, πολλά, πολλοί δείχνουν το δάχτυλο και λένε τι θα πρέπει να κάνετε, τι θα πρέπει να αποφύγετε. Δεν θέλουμε τέτοια πράγματα. Δεν θέλουμε να διχάζουμε τους κλάδους ή να τους κατακαιρματίζουμε, ιδιαίτερα στη γεωργία. Θα ήθελα να πω με σαφήνεια το εξή. Οι αγρότε γνωρίζουν ότι θα πρέπει να αναλυφθεί η δράση, αλλά αν του περιθωριοποιούμε, του τριμώχουμε σε μια γωνία και του λένε ότι αυτοί δημιουργούν το πρόβλημα, όχι, λάθο, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο πώ μιλάμε. Και οι ε, γεωργοί βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση. Είναι ανήμποροι, δεν έχουν ε, σωστή πηξίδα, σωστή κατεύθυνση. Επίσης έχουμε την ε, γεωργία ακριβίας, τη γεωργία συντήρησης. Συμφωνούμε ότι θέλουμε μια πιο φιλοβε φιλοπεριβαλλοντική αγροτική πολιτική. Αλλά θα πρέπει να δώσουμε ξεκάθαρα σήματα και να επιβραβεύσουμε εκείνους που παρέχουν και προσφέρουν έργο και έχουν αποτελέσματα. Έχουμε κάποια στατιστικά. 70% του Παγκόσμιου Γεωργία ελέγχεται από τρει εταιρείε. 90% του παγκόσμιου εμπορίου από τέσσερι εταιρείε και σε ε, οι βασικότεροι, ε, οι περισσότερες αλυσίδες διανομής καρπώνονται το 60% της ε, αγοράς τροφίμων. Θα πρέπει λοιπόν αυτά τα στοιχεία να τα λάβουμε υπόψη πριν αποφασίσουμε να αντιμετωπίσουμε τις κλιματικές αλλαγές. Ευχαριστώ κυρία Μποναφέ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Συνάδελφοι, ότι υπάρχει σήμερα κλιματική και κατεπέγουσα αλλαγή, ανάγκη είναι κάτι το οποίο πρέπει να το πάρουμε πολύ σοβαρά και φυσικά ακόμα και εδώ. Η άνοδο τη Δημοκρασία δείχνει ότι τα τελευταία 50 χρόνια υπάρχει τάση αύξηση χωρί προηγούμενο. Κάθε Ευρωπαίο πολίτη έχει πλέον ε, ζήσει κάτι ανάλογο, ε, έκτακτα καιρικά φαινόμενα, πολλέ φορέ είναι και καταστροφικά. Και ταυτόχρονα αυξάνεται και η δημογραφική πίεση στον πλανήτη. Ήμασταν το 2 ε, δισεκατομμύρια και τώρα είμαστε 7 και θα φτάσουμε μέχρι το 2050 10 δι. Εάν θέλουμε λοιπόν να προστατεύσουμε τον πλανήτη και την ποιότητα ζωή των μελλοντικών γενεών, πρέπει να αλλάξουμε το μοντέλο τη ανάπτυξη σήμερα. Και θα πρέπει να δράσουμε για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, εφαρμόζοντα πολιτικέ σε όλου του τομεί. ε, μηδενός εξαιρουμένου. Θα πρέπει καταρχάς να προστατεύσουμε αυτό που παράγουμε, προστατεύοντα και το περιβάλλον και τη βιοπικιλότητα. Και μαζί σκέφτομαι και την καθαρότερη ενέργεια, την βιωσιμότερη γεωργία, το μεγάλο θέμα τη κινητικότητα μέσα μεταφορά τα οποία είναι λιγότερο ρηπογόνα και αποτελεσματικά. Πρέπει να βρούμε νέα μοντέλα της κοινή της ε, μικτής ε, μεταφοράς με νέες επαγγελματικές δεξιότητες, με καινοτομία και προγράμματα για αλλαγή στο σύστημα κατανάλωσης, με κυκλική οικονομία και νέες δυνατότητες για την μετατροπή των αποβλήτων και τη διαχείρισή τους, να χρησιμοποιούνται αντί για, τα, για τις πρώτες ύλες. Είναι ένα σημαντικό θέμα η απασχόληση και η εργασία. Πρέπει να σκεφτούμε τα νέα επαγγελματικά επαγγέλματα και πρέπει να μην αυταπατώμεθα. Θέλουμε μια θετική πορεία. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε χωρί του ε, κατάλληλου πόρου και να κάνουμε ότι τίποτα δεν συνέβη. Δεν θα πετύχουμε τίποτα. Οι στόχοι τη κυρία Ursula von der Leyen ωραίοι είναι, αλλά πρέπει να χρηματοδοτηθούν. Ε, θα πρέπει λοιπόν να έχουμε και φιλοδοξότερη πρικοδότηση ε, των προγραμμάτων αυτών για να πετύχουμε του κλιματικού μα στόχου. Θα πρέπει να δούμε νέα προγράμματα, γιατί αλλιώ θα χρειαστεί να βρούμε νέου πλανήτε για να κατοικήσουμε. Και θα πρέπει πρέπει αντί να χρηματοδοτούμε τέτοια ερευνητικά προγράμματα να κοιτάξουμε τον όμορ... Ε, πανέμορφο αυτό πλανήτη μα να τον φροντίσουμε. Όχι μόνο γιατί μα το ζητάει η Γκρέτα, αλλά γιατί θέλουμε να προστατεύσουμε και να τη φυλάξουμε το δικό μα μέλλον. Ευχαριστούμε για ένα λεπτό ο κύριος Στεφανούτσα. Ευχαριστώ. Κάθε φορά που συζητούμε τις κλιματικές αλλαγές σε αυτό το σώμα, κοιτάζω εκεί στο θεωρείο, τους νέους. Γιατί εκεί, για εκείνους μιλάμε. Θέλω λοιπόν να σας μεταφέρω ένα μήνυμα σήμερα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας γίγαντας για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ταυτόχρονα και ένας νάνος ό,τι αφορά την προσαρμογή της στις ε, ανάγκες των, που απαιτούν οι κλιματικές αλλαγές. Εδώ λοιπόν πρέπει να προσαρμοστούμε ευθύ αμέσω. Πρέπει να προσαρμοστούμε σε, στις κλιματικές αλλαγές με τον τρόπο που οικοδομούμε τα σπίτια μας, ε, πώς αντιμετωπίζουμε την κλιματική μετανάστευση και πώς τις πλημμύρες, πώς προβλέπουμε τις πυρκαγιέ και τι αντιμετωπίζουμε, πώ φτιάχνουμε καλύτερε στέγε ηλιακέ τη πόλη μα. Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ αναχέτηση, προσαρμογή και μετανάστευση. Στη Γαλλία, η μόνωση των σπιτιών με την ε, αντιμετώπιση των αερίων, εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου τελικά καταλήγει να είναι μετριασμό των κλιματικών αλλαγών. Αλλά μόνο το 3% των επενδύσεων μα, ε, όπω υπολογίζεται στο ε, δημοσιονομικό πλαίσιο, το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο, υπολογίζει χειρίζεται έτσι ως ε, μέσο για την προσαρμογή και τον αταιασμό. Ευχαριστούμε για ένα λεπτό κύριο Μπλό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Έχουμε να κάνουμε με μια τεράστια καταστροφή, αλλά διπλή. Η μία είναι αποτέλεσμα ε, δικής μας ε, ε, Και για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες εκατομμύρια άτομα κατέβηκαν στου δρόμου της Ευρώπη. Ευχαριστούμε όλα τα άτομα που κατεβαίνουν στον δρόμο και μα καλούν να σεβαστούμε την επιστήμη. Και είναι σαφέ το μήνυμα. Δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί η παρούσα κατάσταση. Αλλά μέχρι στιγμή για την κλιματική προστασία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έχει μόνο ευχολόγια και 5,5 δισεκατομμύρια πηγαίνουν σε προγράμμα για το φυσικό αέριο. Και δυστυχώ στη Γερμανία είναι ευχολόγια και αυτά που επιχειρούνται μέχρι τώρα. Ωραίο που οι σοδημοκράτε ε, ζήτησαν να γίνει μια συζήτηση για το θέμα αυτό. Αλλά δεν αρκεί το να συζητάμε. Θέλουμε επιτέλους ε, πράξη. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Λίμα. Εδώ έχουμε διάφορους νευρωτικούς που μιλάνε συνεχώς για μια κλιματική καταστροφή και λένε ότι υπάρχει πολύ διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρά μας. Και ε, κυρίως τα τελευταία 150 χρόνια και για ένα πολύ λογικό λόγο. Αν δείτε την ιστορία της υδρογείου θα δείτε ότι και σε παλιότερες εποχές είχαμε πολύ υψηλότερο ποσοστό ενώ τώρα έχουμε μόνο 400 ppm και δεν υπάρχει κανένας συσχετισμό μεταξύ πυκνότητας διοξιδίου του άνθρακα και ε, κλίματος. Υπάρχουν στερικές φωνές ότι αν ανεβούμε κατά 100 ε, ε, μέρη ανά εκατομμύριο θα ανέβει η θερμοκρασία κατά 2 βαθμούς. Αυτό σημαίνει ότι αν την εποχή των δεινοσαύρων που είχαμε 2.000 μέρη ανά εκατομμύριο, δηλαδή 1.600 παραπάνω από τώρα, η θερμοκρασία θα έπρεπε να είναι 32 βαθμούς παραπάνω. Και θα ήταν περίπου στους 50 ή και παραπάνω. Πολλά στοιχεία αυτό είναι δύσκολο να τα καταλάβει ο α ή ο β πολιτικός. Η κλιματική αλλαγή είναι ο κανόνας, όχι η εξαίρεση. Καλό θα ήταν να, προσαρμο... να προσαρμοζόμαστε στην αλλαγή του κλίμακος. Η μάχη αυτών των δών κυχωτών ε, κατά του κλίματος μπορεί μόνο να χαθεί. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Τέρτ, ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να δούμε τι κάνουμε. Γιατί όλοι μιλάνε για επιστήμη. Αλλά ορισμένοι μιλάνε σαν να είναι μαγεία όλα αυτά. Πολύ ιδεολογικές προσεγγίσεις. Δεν ε, χρησιμοποιούμε την κοινή λογική. Κάθε φορά χρησιμοποιούμε και πιο ακραίο λεξιλόγιο. Και ε, απομακρυνόμαστε από τη λογική και πηγαίνουμε σε πολύ ακραίες θέσεις. Αυτός ο τίτλος ε, «Κλιματική επίγουσα κατάσταση». Όλα αυτά βασίζονται σε ιδεολογήματα. Και έχουμε και αυτούς τους νέους ε, κληρικούς που θέλουν να αποκλείσουν ή ουσδήποτε αναρωτιούνται αν είναι σωστά όλα αυτά ή έχουν διαφορετικές θέσεις. Πιστεύω ότι όλοι πρέπει να κάνουμε προσπάθεια για να μην επιτρέψουμε αυτή η φανατική, η φανατική τρελή παπά